καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και ένα μεγάλο τμήμα των νομοθετικών εργασιών του Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή Περιβάλλοντο θέλει πολύ να προστατεύσει τι συνθήκε για την υγεία, την ισότητα τη πρόσβαση στην περίθαλψη για όλου του ασθενεί στην Ευρώπη και για τα μέγιστα επίπεδα ασφαλεία σε όλη την επισητιστική, στην, ε, αλυσίδα των τροφίμων. Είναι καρδιοχειρούργο Αντρικάτη, έχει 20 χρόνια εμπειρία στον ιατρικό του τομέα στη Λιθουανία ήταν Υπουργό ε, Υγεία από το 2012 μέχρι το 2014, περίοδο κατά την οποία η Λιθουανία είχε και την ε, Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω από, μετά τα 20 χρόνια κοινοβουλευτικής ε, εμπειρίας, διότι ήταν βουλευτής για 6 θητείες στο Λιθουανικό Κοινοβούλιο, πρόσθεσε και αυτή την εμπειρία, ήταν και πρόεδρος της Επιτροπής για Ευρωπαϊκά Θέματα και ηγήθηκε της Λιθουανικής Αντιπροσωπείας για τη Σύμβαση για το Μέλλον της Ευρώπης. Όπως γνωρίζετε αυτή η ακρόαση διοργανώνεται από την Επιτροπή Περιβάλλοντος σαν καθήλυνα αρμόδια επιτροπή και την Επιτροπή Γεωργίας ε, που είναι συνδεμένη επιτροπή. Έχουμε 45 ομιλητές και 6 από την Επιτροπή Γεωργίας. Να υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με τις κατακτήριες γραμμές για την έγκριση των υποψηφίων Επιτρόπων αξιολογεί τους υποψήφιους επιτρόπους στο Κοινοβούλιο βάσει των γενικών τους ικανοτήτων, την αφοσίωσή του για τα ευρωπαϊκά θέματα και την ε, προσωπική του ανεξαρτησία επαληθεύει κατά πόσο γνωρίζουν τα συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια και τη δυνατότητα που έχουν όσον αφορά την επικοινωνία. Πριν από την ακρόαση, ο Επίτροπος απάντησε γραπτός στις ε, γραπτές ερωτήσεις που του θέσαμε οι απαντήσει στα αγγλικά διανεμήθησαν στου βουλευτέ στι 26 Σεπτεμβρίου και όλε οι άλλε γλωσσικέ εκδοχέ έχουν διανεμηθεί χτε το απόγευμα. Όσον αφορά τη δομή τη συζητήσεω, ο υποψήφιο επίτροπος θα κληθεί να προβεί σε μια εισαγωγική δήλωση που δεν θα κρατήσει πάνω από 10 λεπτά και μετά στο τέλος της συνεδριάσεως θα έχει ένα πεντάλεπτο στη θέση του τόσο ώστε να προβεί σε μια σύνοψη, σε καταληκτική δήλωση. Θα υπάρξει χρόνο για 45 ερωτήσει βουλευτών κατά τη διάρκεια τη ακρόαση. Σε τέσσερι ομάδε θα μοιραστούν ερωτήσει. Η πρώτη ομάδα θα αποτελείται από 7 μεγαλύτερε ερωτήσει, 5 λεπτού, με το σύστημα ping-pong που θα ακολουθήσουμε. Θα τεθούν ερωτήσει εκπροσώπου των πολιτικών ομάδων. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα έχουμε ένα λεπτό για την ερώτηση, δύο λεπτά για την απάντηση, ένα λεπτό για συμπληρωματική ερώτηση και ένα λεπτό για συμπληρωματική απάντηση. Μετά θα υπάρξει δεύτερος γύρος, 26 συντόμων ερωτήσεων, τριών λεπτών συνολικά, που θα τεθούν από τα μέλη της Επιτροπής ΕΜΒΗ. Σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε ένα λεπτό για την αρχική ερώτηση, δύο λεπτά για την απάντηση. Και στον τρίτο γύρο όμως έχουμε συμπεριλάβει τις ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής Γεωργίας Ερωτήσεις σύντομες θα είναι αυτές και θα καταλήξουμε με 7 σύντομες ε, ερωτήσεις από την πλευρά των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Το τέλος λοιπόν για, μάλλον, για να ολοκληρώσουμε τη συνεδρίαση εγκαίρω, διότι προβλέπει να, θα πρέπει να διαρκέσει ακρόαση τρει ώρε για να είμαστε εγκαιροί καλούμε και του συναδέλφου στον υποψήφιο επίτροπο να σεβαστούν το χρόνο ομιλία. Θα υπάρξουν 5 δευτερόλεπτα ανοχής για του βουλευτέ και 10 δευτερόλεπτα ανοχή για τον επίτροπο. Αν περάσουν αυτά, το μικρόφωνο θα κλείνει. Ένα αστερίσκο θα εμφανίζεται επί τη οθόνη 10, λεπτά, 10 συγγνώμη, δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του χρόνου ομιλία και το σφυράκι του Προέδρου πάση περιπτώσει θα υπενθυμίζει ότι λύγει ο χρόνος. Υπενθυμίζω ότι η διαρμηνία προβλέπεται σε 23 γλώσσες. Συνεπώς όλοι οι ομιλητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα τους. Η συζήτηση επίσης μεταδίδεται και στο διαδίκτυο μέσω streaming στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου και από εκεί θα μπορείτε να κατεβάσετε την ηχογράφηση της ακρόασης. Δίνω αμέσω το λόγο στον υποψήφιο επίτροπο, τον κύριο Ανδρουκάητης, ούτως ώστε να προβεί στην αρχική του δήλωση. Έχετε το λόγο.